Συνεχίζουμε τις ψηφοφορίες. Έχετε την ηλεκτρονική σας κάρτα όλοι, φαντάζομαι. Παρακαλώ, δοκιμάστε τι αν δουλεύει για να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Λοιπόν, τροποποίηση του κανονισμού 2371 κάθετος 2002 του Συμβουλίου Διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλληλευτικών πόρων στο πλαίσιο της ΚΑΛΠ. Εισηγητής ο κύριος Χάτστον. Έτοιμοι, μπορούμε να αρχίσουμε. Αρχίζουμε λοιπόν. Στην νομοθετική πρόταση δεν έχουμε τροπολογίες. Ε, συγγνώμη, νομοθετική πρόταση έτσι όπως τροπολογήθηκε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη η ψηφοφορία. Χωριστή ψηφοφορία για την παράγραφο 2 του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος. Αρχή απορρίπτεται. Χωριστή ψηφοφορία της παραγράφου 3. Αρχίζει ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος. Αρχίζει. Ολοκληρώνεται, εγκρίνεται ομόφωνα. Το επόμενο θέμα μας είναι η διατήρηση των αλλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νερών θαλάσσιων οργανισμών. Αρχίζουμε με την τροπολογία 22. Αρχίζει ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Αρχίζουμε. Κλείνει ψηφοφορία. Εγκλίνεται. Τροπολογία 5. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Αρχίζει. Ολοκληρώνεται. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Αρχίζει. Ολοκληρώνεται. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Αρχίζει, ολοκληρώνεται, απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Αρχίζει, λίγη, εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Αρχίζει, λίγη, εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Αρχίζει. Ολοκληρώνεται. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. 32. Ναι. Αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 11, 33. Αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1. Αρχίζει, κλείνει, Εγκρίνεται. Καταπίπτει η 12. 35. Αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 13. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος. Πρώτα. Αρχίζει. Κλείνει εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος αρχίζει, κλείνει, απορρίπτεται το δεύτερο μέρος. 37 αρχίζει, κλείνει, απορρίπτεται. 38 αρχίζει, κλείνει, απορρίπτεται. 15 Αρχίζει, κλείνει. Εγκρίνεται. Τριάντα εννέα. Αρχίζει. Όχι. Συγγνώμη. Δεκάξι. Αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. 40. Αρχίζει. Κρίλιν εγκρίνεται. 41. Αρχίζει. κλείνει, συγγνώμη, εγκρίνεται. 43. Αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. 44. Αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. 17. Αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. 18. Αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. 45. Αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 47. Αρχίζει, κλείνει. Εγκρίνεται. Αριθμός ένα, Αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. 20. Αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. πίπτη 2. Και φτάνουμε στην ε, νομοθετική πρόταση έτσι όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει, κλείνει, εγκρίνεται και τώρα στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Αρχίζει, κλείνει, εγκρίνεται, ομόφωνα. Συγχαρητήρια κύριε Χάφτον. Κύριε Γκάλαχερ. Η κυρία Φράγκα. Μία ερώτηση στην Κομισιόν, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα αυτό. Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής, εγκρίθηκε η έκθεση, εάν την πρόταση αυτή θα την εγκρίνει η Κομισιόν στον κανονισμό για τη Μαύρη Θάλασσα, θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν εδώ να μπορεί να απαντήσει. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ε, uh, Μέρος της Κομισιόν. Υποστηρίζουμε την ε, συμπερίληψη και της Μαύρης Θάλασσας. Είχαμε συζητήσεις και με τους Αρμενίους και με τους ε, Βουλγάρους. Καταρχήν λοιπόν ναι, μπορώ να απαντήσω. Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Αναθέτουμε στον κύριο Γκάλαχερ να κάνει την διαπραγμάτευση του θέματος αυτός. Σε σχέση με αυτό το θέμα υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Εάν όχι, περνούμε στο επόμενο. Το 5. Ε, πρόεδρε, εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία της παρουσίας ε, της Κομισιόν για να τη ρωτήσω. Και όλοι μας την αντιπροσωπεία πριν από μερικές μέρες σε διεθνή ύδατα, επαναλαμβάνω σε διεθνή ύδατα, όπου υπήρξαν ζητήματα μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης. Συλληφθήκαν δύο αλληλευτικά Ιταλικά τα οποία παραμένουν συλληφθέντα στη Λιβύη. Είναι ένα αίτημα που εδώ και χρόνια, με το οποίο υπάρχει και εδώ, εδώ και χρόνια πρόβλημα και επαναλαμβάνω στην Κομισιόν, ε, συνλήφθησαν δύο αλλιευτικά Ιταλικά σε διεθνή ύδατα από τη Λιβύη και θα ήθελα οι βουλευτές εδώ να το συζητήσουμε αυτό στην επόμενη συνεδρίαση για τη Μεσόγειο. Ε, αναμένω την απάντηση της Κομισιόν. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν μπορεί να απαντήσει αυτό το θέμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Προηγουμένως έδωσα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι αφορούσε ένα θέμα, ένα ερώτημα του θέματος που συζητούσαμε. Τώρα για κάτι άλλο το οποίο δεν προβλέπεται και μπορεί να τεθεί διαφορετικά, δεν ξέρω. Εάν μπορεί να απαντήσει η Κομισιόν και θέλει, έχει καλώς. Διαφορετικά, Τι να πω, η Κομισιόν δεν έχει κανένα λόγο να είναι προετοιμασμένη και ενήμερη για να απαντήσει σε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Μπας περιπτώσει. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε, αλλά δεν συμφωνώ μαζί σα. Οι Λίβοι δεν μας ειδοποίησαν ότι θα συλλάμβαναν αυτά τα δύο αλλιευτικά σε διεθνή υδάτα. Είναι μία πράξη που επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια. Η Κομισιόν θα έπρεπε να έχει κάποια εικόνα, διότι αυτή η ιστορία δεν έχει τέλος. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να προετοιμάσουμε έκθεση για ε, ένα τέτοιο γεγονός το οποίο είναι τόσο σοβαρό και το οποίο έχει τέτοια έκθεση και επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια. Βεβαίω και δεν μας προειδοποιούν όταν θα γίνει τέτοιου είδου πειρατεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εάν είναι προετοιμασμένη η Κομισιό, έχει καλώ. Ούτε προβλέπεται, ούτε ίσω είναι και η κατάλληλη στιγμή. Νομίζω ότι εγώ με πολύ καλή θέληση και θετικό πνεύμα Σα άφησα μιλήσει. Τώρα, αν θέλει να απαντήσει η Επιτροπή ή δεν μπορεί να απαντήσει, προφανώ δεν μπορούμε να την υποχρεώσουμε. Υπάρχουν διαδικασίες που προβλέπουν κάτι τέτοιο και σίγουρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δέουσες διαδικασίες. Θέλει η Κομισιόν να απαντήσει στο ερώτημά σας? Εάν όχι, περνούμε στο επόμενο θέμα. Το σημείο 5. τροποποίηση του κανονισμού 1098 του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολιτού σχεδίου τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής και για τις αλληλευτικέ δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων. Η Επιτροπή είχε παρουσιάσει το θέμα αυτό την 21η Ιουνίου. Δίνω αμέσω τώρα το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Βρίσκομαι εδώ σήμερα ε, συζητάμε σήμερα την τροπολογία για τα συμπερασμάτα του Συμβουλίου για το ετήσιο, ε, για το πολιτέ σχέδιο για τα θέματα γάδου της Βαλτικής. Αυτός ο κανονισμός χρειάζεται να τροποποιηθεί διότι όλοι οι κανονισμοί πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τη συνθήκη της Λισαβόνας η Γραμματεία πρότεινε να προχωρήσουμε με αυτές τις ε, τροπολογίες και βασικά έχω ακολουθήσει την πολιτική που έχει ακολουθήσει η πολιτική μας στο παρελθόν. Αυτός ο κανονισμός υπάρχει εδώ και πέντε χρόνια και έχουμε παρατηρήσει ότι δεν λειτουργεί όπως θα θέλαμε. Η Κομισιόν προτείνει να μην κάνουμε απλά ε, τις συνήθειες τροπολογίες προσαρμογής του κανονισμού στη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά πρέπει να πάμε πιο πέρα. Ε, διότι αυτός ο κανονισμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σε αυτό που συμβαίνει για τα αποθέματα γάδου. Και αυτό δηλώθηκε, δηλώθηκε σαφώς πέρυσι από το ESTF. Αυτοί είναι οι λόγοι λοιπόν για τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. τα αποθέματα γάδου βρίσκονται σε καλύτερη θέση τώρα χάρη στο πολιτέ σχέδιο, αλλά το πολιτέ σχέδιο δεν είναι αρκετά ευέλικτο. Πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να θέσουμε ως στόχο να εισάγουμε περισσότερη ευελιξία στον κανονισμό. Γι' αυτό ήθελα να σας μιλήσω σήμερα. Ε, λάβαμε μια σειρά συστάσεων από το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την ε, Βαλτική. Θα ήθελαν και αυτοί περισσότερη ευελιξία. Βάσει φυσικά επιστημονικών συμβουλών. Αυτή είναι η επιστημονική εκθέση που ανέφερα νωρίτερα. Βάσει αυτή τη εκθέση θα προτείνει τροπολογίε η Κομισιόν, αλλά ακόμη δεν έχουμε λάβει τίποτα γραπτό. Η Κομισιόν έχει προτείνει να υπάρχει ένα σχέδιο διαχείρισης πολλών ειδών, πολλαπλών ειδών και αυτή τη στιγμή αυτό βρίσκεται υπό μελέτη. Το σχέδιο λοιπόν για το γάδο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και την κατάσταση των υπόλοιπων ειδών. Καταλαβαίνω ότι η δημιουργία ε, κατά τη τέτοιου σχεδίου προγράμματος θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό αλλά ευτυχώ, σύμφωνα με τι πληροφορίε που έλαβα εγώ και ίσω θα μπορούσε να το επιβεβαιώσει η Κομισιόν, αυτό το πρόγραμμα, το σχέδιο θα ε, παρουσιαστεί λίγο με κάποια καθυστέρηση σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Χρειαζόμαστε νέα επιστημονικά στοιχεία αυτό το αρκετά ευρύ σχέδιο ευρύες εφαρμογής πρέπει να συσταθεί σωστά. Αλλά χρειαζόμαστε αρχικά ένα καλό σχέδιο για το απόθεμα γάδου. Μπορούμε να βελτιώσουμε κάπως το υπάρχον πολιτές σχέδιο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε μια μερική εισαγωγή του ε, σχεδίου διαχείρισης πολωνιδών πολλών αποθεμάτων. Προτείνω λοιπόν να λάβουμε υπόψη τη θνησιμότητα των ψαριών στα αποθέματα που υπάρχουν. Θα μπορούσαμε ίσως να αυξήσουμε λίγο τη θνησιμότητα αυτού του αποθέματος. Γίνεται εκτενής ανάλυση του κειμένου αυτή τη στιγμή. Έχουμε 1,3 ως θνησιμότητα και βάσει του το τρέχον σχέδιο δεν περιλαμβάνει κάποιο είδου μηχανισμό αύξηση του αριθμού αλληλευτικών ημερών. Δηλαδή των ημερών που ε, εκτός λιμένος. Αυτή είναι η τροπολογία 9 που προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Επίσης μικρότερα αλληλευτικά σκάφη ε, μήκους χαμηλότερο των 12 μέτρων. Θα πρέπει να επιτρέπεται να ψαρεύουν ε, εντός 12 μιλίων από τις ακτές. Εδώ μιλάμε για τους καλοκαιρινούς μήνες. Ε, αυτή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει λογικά να επηρεάσει καθόλου το ρυθμό τοκίας και αναπαραγωγής. Διότι περισσότεροι νεαροί οργανισμοί βρίσκονται σε μεγάλο βάθος ε, και εδώ μιλάμε περισσότερο για ε, παράκτια αλληλεία. Επίσης υπάρχουν διατάξεις που αναφέρουν ότι είναι σημαντικό για την επιτυχία του σχεδίου τα κράτη-μέλη να μπορούν να παρακολουθούν την όλη διαδικασία και τα μέγιστα επιτρεπόμενα λίευματα. Είναι σημαντικό πιστεύω να θυμόμαστε τις περιόδους απαγόρευσης της αλίας. Αν και αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό, διότι τα αποθέματα γάδου φαίνονται αρκετά καλά. Υπάρχουν λοιπόν δύο μηχανισμοί που θα μας βοηθούσαν σε για περισσότερη ευελιξία. Στην πρόταση της Κομισιόν λέει ότι οι εκτελεστικές εξουσίες της Κομισιόν πρέπει να ορίζονται καθαρά ε, είτε μέσω κατεξοδότηση πράξεων είτε μέσω εκτελεστικών πράξεων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ταξινόμηση μεταξύ των διαφορετικών διατάξεων. Ε, αυτό καλύπτει σε μια σειρά άρθρων ε, που θα πρέπει να προσαρμοστούν στη συνθήκη της Λεβόνας. Το άρθρο 26 αφορά την υλοποίηση, την εφαρμογή του σχεδίου. Το άρθρο 27 καλύπτει την θνησιμότητα των ηχθείων. Η Κομισιόν λοιπόν τώρα θα ήθελε κατεξουδότηση πράξης για αυτά τα θέματα. Αυτό υποτίθεται, αυτές υποτίθεται θα καλύπτουν τα μη ουσιώδη στοιχεία. Ωστόσο δεν συμφωνώ μαζί τους. Η θνησιμότητα των ψαριών αποτελεί κλειδί για αυτό το πολιτικό σχέδιο. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να εντάσσεται στην κατηγορία των θεμάτων που εξετάζονται με εκτελεστικέ πράξει. Ε, μπορώ να σα προτείνω και άλλε μικρέ αλλαγέ. Έχουμε διατάξει στο κείμενο τη Κομισιόν που επιτρέπουν ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκεί εξουσίε δύναμη της τροπολογίας 12. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. Αυτά είχα να πω μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαλένσα. Και ε, από τα τέσσερα άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο, το πρώτο άτομο που θα μιλήσει είναι ο κύριος Στραβέλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαλέσα για την εκθεσή του. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα για τα οποία δεν συμμερίζομαι την άποψή σας. Όταν εξεταζούμε το αποθέματα γάδου στη Βαλτική, ουσιαστικά αυτό αποτελεί διπλό κίνδυνο από νομική άποψη. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια πολύ σοβαρή διαδικασία αφαλάτωσης στη Βαλτική. Ειδικότερα ο γάδος εξαρτάται ιδιαίτερα από την αλατότητα των υδάτων. Αυτό που βλέπουμε εμείς ε, να συμβαίνει είναι ότι η γάδη είναι περίπου 35 εκατοστών και δεν είναι καλές οι συνθήκες για αυτούς παρότι είναι περισσότεροι. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο αισθάνονται περίεργα τα ψάρια αυτά, ίσως ε, λόγω της αφαλάτωσης. Γνωρίζουμε όμως επίσης, ε, γι' αυτό δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, γνωρίζουμε όμως ότι και η αναπαραγωγή, η οτοκία μάλλον των γάδων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στα βαθύτερα ύδατα της Βαλτικής. Αλλά τι έχουμε στα βαθύτερα ύδατα της Βαλτικής, έχουμε νεκρό βυθό τεράστιες δηλαδή επιφάνειες χωρίς ε, στοιχεία διατροφικά που αναγκάζουν τους γάδους να ανεβαίνουν σε μικρότερο βάθος όπου δεν αισθάνονται άνετα. Όπου δεν ε, μπορούν να διατηρήσουν την καλή τους κατάσταση. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά το γάδο στη Βαλτική από ότι είναι αποδεκτό. Θεωρώ λοιπόν ότι οι τροπολογίες 4, 5, 9 και 10 είναι λίγο υπερβολικά αισιόδοξε. Ε, καλό είναι να είναι κανείς αισιόδοξος, αλλά όχι τόσο πολύ. Πιστεύω ότι θα ήταν σοφό να αναμένουμε να δούμε το σχέδιο για τα πολλαπλά είδη. Καταλαβαίνω ότι οι σημαντικές παρατηρήσεις ε, του κ. Βαλέσα όσον αφορά το σχέδιο πολλαπλών ειδών. Φυσικά πρόκειται να καθυστερήσει τότε. Θα αντιμετωπίσουμε διπλό κίνδυνο. Το κατανοώ αυτό. Αυτά είχα να πω εγώ για σήμερα. Μάλλον για αυτή τη φορά που μιλάω ο κύριος Τόρβαλτς. Ευχαριστούμε τον κύριο Τόρβαλτς και τώρα ο κ. Κρίστιανσον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Σιγητή για το σχέδιο που μας παρουσίασε, το σχέδιο έκθεσης. Θα πρέπει να προσέξουμε τις συνέπειες σε περίπτωση προσαρμογής αυτής της νομοθετικής πράξης στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, το θέμα εδώ είναι πολιτικό. Όπως ανέφερε ο εισηγητής ε, στην τροπολογία 4 με τους ε, στόχους θνησιμότητας των νυχθείων, Πρώτα απ' όλα, επειδή αυτή τη στιγμή ε, πραγματοποιούμε ανάλυση επακόλουθων, όπως ανέφερε και ο κύριος Τόρβαλτς ε, στις ανοιχτές θάλασσες και στο STCF, και θέλω να περιμένω τα αποτελέσματα αυτών πριν προβούμε σε περαιτέρω προσαρμογές. Θέλω φυσικά ένα μακροπρόθεσμο αηφόρο αλλά και ρεαλιστικό σχέδιο για την αλία του γάδου στη Βαλτική. Έτσι λοιπόν οι πολιτικές αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις με συνέπειες για τον γάδο στη Βαλτική θα πρέπει να αναμένουν τα αποτελέσματα των εν λόγω μελετών. Δεν χρειαζόμαστε άμεσες αντιδράσεις και βραχυπρόθεσμες λύσεις το χρωστάμε στη βιομηχανία να τους ε, δώσουμε, να τους προσφέρουμε μια μακροπρόθεσμη νομοθεσία για πολλά έτη. Διαχειριζόμασταν την αλία γάδου στη Βαλτική με λανθασμένο τρόπο. Αυτό δεν συμφέρει κανέναν. Και δεν συμφέρει κανέναν να συνεχίσουμε να ψαρεύουμε γάδο στη Βαλτική με τρόπο μη βιώσιμο. Εάν τα αποθέματα γάδου βελτιώνονται, Εξακολου... Παρότι τα αποθέματα βελτιώνονται, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε ένα καλό σχέδιο διαχείριση. Οπότε ας προσαρμόσουμε την νομοθεσία έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση περί της διαχείρισης της αλληλεία σε αυτή την περιοχή. Ήθελα επίση να ρωτήσω την Κομισιόν πού βρισκόμαστε με αυτό το πολιτικό σχέδιο και πότε μπορούμε να αναμένουμε μια πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμένουμε με λοιπόν, υπομονησία να... καλή συνεργασία με τον κύριο Σιγητή. Η κυρία Λεβίν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Συγητή για όλη τη δουλειά που έχει κάνει. Συμφωνώ με όσα είπαν ο κύριος Τόρβαλτς και ο κύριος Κρίστινσαν. Έχουμε ένα σχέδιο μακροπρόθεσμο για το γαδό στη Βαλτική και αυτό επέτρεψε την αύξηση των αποθεμάτων. Αυτό πρέπει να μας χαροποιεί. Παρότι παραμένουν πολλές ανησυχίες όσον αφορά την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των διαφορών ειδών. Παρευρέθη σε ένα σεμινάριο πριν από δύο εβδομάδες για τα οικοσυστήματα που διοργανώθηκε από ένα περιφερειακό συμβουλευτικό ε, γνωμοδοτικό συμβούλιο και συζητήσαμε τα αποθέματα και άλλων ειδών. Εκεί βρίσκονταν αλληλείς που ανησυχούσαν για τα αποθέματα γάδου οι Ελλείς δεν λένε ποτέ έχουμε υπερβολικά πολύ γάδο. Υπάρχουν ε, μεγάλοι πληθυσμοί κοντά στην Πολωνία, αλλά αυτό δεν ισχύει στη Νότια Σουηδία και ακόμη λιγότερο στη Βόρεια Σουηδία. Καλό θα ήταν λοιπόν να, τα αποθέματα γάδου να είναι καλύτερα κατανεμημένα και ελπίζω να υπάρξει μια προσέγγιση ε, πολλαπλών ειδών από την Κομισιόν και αυτή η προσέγγιση να κάνει τη διαφορά. Ελπίζω να είναι αυτό ένα από του στόχου του. Όλοι θυμόμαστε φυσικά τα καταπληκτικά έτη για το γάδο τη δεκαετία του 80. Γνωρίζουμε ότι η Βαλτική θάλασσα έχει τεράστιε δυνατότητε αύξηση των αποθεμάτων, πολύ πέρα από αυτά που αναφέρονται σήμερα. Ε, κύριε Βαλέσσα, αναφέρατε την ιδέα της αυξημένης νησιμότητας ε, στα δυτικά και στα ανατολικά αποθέματα. Αυτό ε, ε, ε είναι αντίθετο με τις συμβουλές της ICC. Πιστεύω ότι το να αυξήσουμε τη θνησιμότητα πάνω από το 1,33 όπως λέει ο κ. Βαλέσα είναι εντελώς λανθασμένη προσέγγιση. Θα δούμε τι θα προτείνει και η Κομισιόν. Έχουν γίνει και άλλε διάφορε προτάσει. Για παράδειγμα, λέμε ότι πρέπει να επιτρέψουμε σε όλα τα σκάφη κάτω των 12 μέτρων να αλλιεύουν κατά την κλειστή καλοκαιρινή περίοδο. Αυτή η περίοδος έχει δημιουργηθεί για να επιτρέπει την αναπαραγωγή των γάδων. Εάν όμως όλα τα σκάφη κάτω των 12 μέτρων μπορούν να αλλιεύουν ελεύθερα εντός 12 μιλιών, πιστεύω ότι αυτή η πρόταση πηγαίνει πολύ μακριά. Αυτό θα έχει συνέπειε. Πιστεύω θα πρέπει να αξιολογήσουμε πολύ καλά αυτέ τι συνέπειε πριν εγκρίνουμε μια τέτοια απόφαση. Δεν ξέρουμε για πόσα σκάφη μιλάμε. Δεν ξέρουμε ποιε θα είναι οι συνέπειε όλου αυτού. Όλα αυτά θα πρέπει να μελετηθούν σωστά σε αυτή την Επιτροπή πριν ε, δώσουμε το ναι σε αυτή την πρόταση. Στην τροπολογία 9 που αφορά την ευελιξία που αναφέρει ο κ. Βαλέσα μιλάνε για αύξηση κατά 10% των ελευθερικών μέρων. Εφόσον δεν αυξήσουμε το, το ποσοστό θνησιμότητας, εάν λάβουμε υπόψη την ιδιαίτερα βέβαια κατάσταση όλων των εκτείων στη Βαλτική. Πιστεύω ότι αυτό θα αντιβαίνει την αρχή της, ε, ε, της αναλογικότητας. Και αυτό, έτσι μας, αυτό με φέρνει στο τελευταίο ερώτημα. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά θα ήθελα να ακούσω τι έχει να πει η Επιτροπή επί αυτού. Στην τροπολογία 2 αλλάζει μια λέξη εκεί, ελάχιστη θνησιμότητα των ψαριών και θα αλλάξει σε ε, θνησιμότητα στόχο. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η αλλαγή. Τι ακριβώς προβλέπει η Κομισιόν εδώ. Ποια είναι η ουσιώδης αλλαγή εδώ. Θα ήθελα πολύ να το καταλάβω. E, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή, τον οποίον ε, συγχαίρω και θέλω να σας πω ότι εδώ ο εισηγητής έχει βασιστεί στις επιστημονικές αποδείξεις. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ότι προφανώς όπως σε κάθε τομέα δεν υπάρχουν ε, επαρκείς επιστημονικές έρευνες και αποδείξεις, ιδίως όσον αφορά τη Βόρειο Θάλασσα, νομίζω ότι εφόσον δεν είναι και ένας τεράστιος χώρος, θα έπρεπε να έχει κανείς επαρκής αποδείξεις, πράγμα το οποίο δεν ευσταθεί. Χρειαζόμαστε ακόμη πολύ περισσότερες. Και γιατί αυτό έχει σημασία, έχει σημασία διότι όπως είπε ένας προλαλήσας πρόκειται ε, για το θέμα π.χ. της αφαλάτωσης που προαναφέρθηκε και δέχεται κατά αυτόν τον τρόπο ο πληθυσμός ε, των αποθεμάτων να μειωθεί. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Τα αποθέματα έχουν ε, αποκατασταθεί και μέχρι στιγμή ε, έχουμε προσάψει στους αλληλείς ότι έχουν κάνει υπερβολική αλίευση αλλά βλέπουμε ότι ενώ είχε μειωθεί η αλληλεία κατά 15% δεν επηρέωσε αυτό τόσο πολύ όσο η αφαλάτωση της βορείου θαλάσσης. Πρέπει λοιπόν να γίνει ένας επακριβής έλεγχος των επιστημονικών αποδείξεων διότι δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο ένας ή ο άλλος παράγων έχει επηρεάσει την κατάσταση ο εισηγητής μιλάει για μία αναθεώρηση του προγράμματος εκμεταλλεύσεως, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Βεβαίως βασιζόμαστε στις επιστημονικές αποδείξεις, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει προσαρμόσει το πρόγραμμα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο κλάδος είναι οριακός όσον αφορά την αποδοτικότητα της εκμετάλλευσης, και ε, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα θετικό, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν, δεν προβλέπει να τροποποιήσει το πρόγραμμα αυτό. Και χωρίς βιώσιμη αλία, όσο και να το συζητάμε, Ίσως ε, θα έπρεπε καλύτερα να μιλήσουμε για τις απορρίψεις, διότι υπάρχουν ακόμη πάρα πολλές απορρίψεις ε, σχετικά ε, με το ψάρι αυτό και δεν έχει αντιμετωπιστεί το θέμα. Η αλληλεία δεν ελέγχεται επαρκώς, διότι σκεφτόμαστε μόνο το συνολικό όγκο των ε, των ε, ψαριών τα οποία ε, έχουν αλλιευθεί χωρίς να μιλάμε για τις απορρίψεις. Το συνέδριο στην Κτίνια που αναφέρατε που απέδειξε ότι ε, τα κράτη ε, της Βορείου Θαλάτης ε, δεν συνεργάζονται βλέπε, απέδειξε πως γίνεται η κατανομή και βάσει ποιων αρχών που βασίζονται σε χερσαία κριτήρια δηλαδή ο κάθε ένας αποφασίζει αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδείγματος χάρη δεν γνωρίζει δεν ξέρει πόσο γίνεται η ενημέρωση δεν γνωρίζει ότι υπάρχει παρανόηση και παραπληροφόρηση και ε, βλέπουμε ότι η βάση της ε, λήψεως αυτών των ε, πληροφοριών λαμβάνονται οι αποφάσεις. Εδώ θα έπρεπε να εναρμονιστεί ο τρόπος ενημέρωσης. Εάν εδώ αναφερθούμε ε, για την ε, ευελιξία σχετικά με τις ημέρες αλίευσης εκτός λιμένου, ε, λιμένος, θεωρώ ότι αυτό είναι καλό, διότι εκεί συνυπολογίζεται και ο καλός καιρός. Βλέπουμε ότι παραδείγματο χάρη σε περίπτωση κακοκαιρίας δεν υπάρχει το ίδιο επίπεδο δυνατοτήτων αλληλείας και υπάρχει πολύ μικρότερο αποτέλεσμα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η ευελεξία είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο και πρέπει να προχωρήσει. Ο κύριος Κιούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Βόρειο Θάλασσα είναι ένα, ένα κλειστός χώρος για αλίευση όπως η Μεσόγειος και ε, είναι κλειστός γύρω γύρω και αποτελείται από διάφορα ψάρια και γι' αυτό εφόσον τονίζουμε το, την αλία του γάδου που είναι ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική τροφή ε, που επιζητείται πάρα πολύ πρέπει να κάνουμε ένα απολογισμό της κατάστασης. Πριν πέντε χρόνια υπήρξαν, ε, υπήρξε μια μεγάλη κρίση και πολλές περικοπές ακόμη και για τα περιφερειακά προγράμματα αλλιεύσης αλλά τώρα έχει συνέλθει και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι βλέπουμε ότι αν υπάρχει υπερβολή η ποσό της γάδου που διατίθεται στην αγορά πέφτει τιμή, αν μειωθεί υπάρχει αύξηση τιμής και γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε ένα management plan. Ε, όταν δούμε όμως πώς έχει εξελιχθεί το πρόγραμμα αλίευσης στην ε, Βόρειο Θάλασσα, έχει σημασία και πώς είναι η περιεκτικότητα της θαλάσσης αυτής σε αλάτι. Και ε, βλέπουμε ότι μέχρι ενός σημείου η κατάσταση είναι απλή όσον αφορά το ποσοστό αλατιού στο νερό, αλλά μετά περιπλέκεται η κατάσταση. Οπότε γι' αυτό πρέπει να έχουμε επαρκή πληροφόρηση για να μπορέσουμε να γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται ε, και ε, να δούμε ότι ε, υπάρχουν ορισμένα τα οποία επηρεάζουν το γάδος ε, διατρέφεται ε, με ε, γόνους, με μικρές ρέγγες και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διατύπωση του προγράμματα διότι βλέπουμε ότι όταν ισχύουν τα τάκ δεν υπάρχει πλέον αλίευση ενώ υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα εάν το ψάρι παραδοθεί στην αγορά φρέσκο αντί να ψηφίζουν δύο-τρεις μέρες και μετά να τρέξουν να τα δώσουν κατευθείαν ε, στις βιομηχανίες. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπήκα σε αυτή, τη σε αυτή τη συζήτηση γιατί πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική. Είμαι βέβαιος ότι οποιαδήποτε γραμμή συζήτησης που ισχυρίζεται ότι δεν έχουμε επαρκή επιστημονικά στοιχεία ουσιαστικά ψεύδεται. Θα σας δώσω δύο-τρία παραδείγματα. Γνωρίζουμε ότι η αλατότητα της Βαλτικής μειώνεται και γνωρίζουμε και γιατί. Πρώτον, βρέχει περισσότερο πάνω από τη Βαλτική. Βρέχει διότι ο Βόρειος ε, Ατλαντικός, ε, η ταλάντωση στο Βόρειο Ατλαντικό βρίσκεται σε άλλη θέση, έχει μετατοπιστεί και αυτό επηρεάζει τις βροχοπτώσεις. Αυτό είναι γεγονός εδώ και 30 χρόνια το να λέμε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε περισσότερες ε, επιστημονικές εκθέσεις γι' αυτό είναι σαν να μην διαβάζουμε αυτά που γνωρίζουμε ήδη. Ο δεύτερος ε, λόγος είναι οι ήπιοι χειμώνες. Γνωρίζουμε ότι το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο έρχεται στη Βαλτική. Για ποιο λόγο, διότι τα βόρεια κομμάτια είναι παγωμένα το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Η πίεση των νερών είναι χαμηλότερη από παλιά και γι' αυτό το λόγο μπορούσαν να μπαίνουν τα ε, θαλάσσια νερά και τώρα δεν παγώνουν πια τα νερά αυτά, το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερη αλατότητα. Διότι τα ρεύματα θαλασσιού δεν εισέρχονται στη Βαλτική επαρκώ το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Εάν αυτό συνεχίσει για 20-30 χρόνια, δεν θα έχουμε πλέον, θα πάψει να υπάρχει γάδο στη Βαλτική, στα νότια μέρη τη Βαλτική, διότι χρειάζεται αλατότητα 11 ο γάδο διαφορετικά δεν τοκί με χαμηλή αλατότητα. Αυτά είναι γεγονότα. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι μεγάλες περιοχές του βυθού της Βαλτικής είναι νεκρές. Και το να λέμε ότι χρειαζόμαστε και περισσότερες έρευνες και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία είναι απλά άρνηση ενός ορατού γεγονότος και αποδεδειγμένου. Και βλέπετε ότι παθιάζομαι με το θέμα και ζητώ συγγνώμη, αλλά εκνευρίζομαι όταν βλέπω να μην κοιτάμε τα πράγματα στα μάτια. Είναι απλά ανόητο. Ευχαριστούμε κύριε Θόρβαλτ. Κύριε Τότς, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κάποιες σύντομες και γενικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, πολλέ από αυτέ τι διαδικασίε ευθυγράμμιση ε, εξετάζονται αυτή τη στιγμή από την παρούσα επιτροπή και θέλω να επαναλάβω αυτό που έχω πει πολλέ φορέ. Χρειάζεται να προχωρήσουμε ω θεσμικά όργανα ώστε να καταλήξουμε κάπου και όχι απλά να τα εξετάζουμε όλα αυτά σε πλαίσιο διαφόρων διαδικασιών Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Δεύτερον, αναγνωρίζει ο εισηγητής κοινά σημεία μεταξύ των διαφόρων αυτών διαδικασιών ευθυγράμμιση. Σε πολλέ από αυτέ τι διαδικασίε η Κομισιόν προσπαθεί να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο και επαναλαμβάνω πράγματα που έχω ήδη πει σε γενικού περιεχομένου συζητήσει όσον αφορά την ευθυγράμμιση για το γάδο τη Ιρλανδική θάλασσα. Είναι ότι τα σχέδια διαχείριση πρέπει να τηρούνται και επίση και εγώ θα κάνω προτάσει που θα πρέπει να ενταχθούν στην πρόταση της Κομισιόν. Το, η τρίτη παρατήρηση αφορά το γεγονό ότι πολλέ από τι προσαρμογέ που προτείνει ο εισηγητή προέρχονται από τον εκνευρισμό λόγω τη αργή απόκριση τη Κομισιόν, που δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα τα οποία εμφανίζουν τα τρέχοντα σχέδια. Και όταν λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα επειδή προσπαθούμε να επιτύχουμε ένα σχέδιο πολλών ειδών, αυτό είναι ένα κομμάτι του προβλήματος, γιατί μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα στο μεταξύ. Απλά η Κομισιόν δεν ασχολείται με αυτές τις τροπολογίες. Πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να μας ακούσει διότι υποψιάζομαι ότι θα το ακούσουν πολλές φορές μέσα στους επόμενους μήνες. Θα ήθελα επίσης να πω ότι όλα αυτά συνοψίζονται σε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν πρέπει να χάνουμε από τα μάτια μας ε, την μεταρρύθμιση της κοινής αλλιευτικής πολιτικής. Δηλαδή ότι ουσιώδης περιφερειοποίηση είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να αντιμετωπίσουμε ζητήματα τέτοιου είδους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά. Ε, βέβαια ε, όλα τα σχόλια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και πρέπει να σας πω ότι μου, ε, μου... με κατηγόρησαν ότι η οι προτάσεις μου ξεπερνούν τα όρια της, ε, του εγγράφου αυτού. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προέβη στις τροποποιήσεις, οπότε εγώ ασχολήθηκα με τις τροπολογίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θέλω να σας πω ότι πρέπει να αντιδράσουμε και στο τι γίνεται ε, στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή, όπου το πρόγραμμα χρειάζεται περισσότερο χρόνο, πρέπει ε, να περιμένουμε, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι ότου διευκρινιστεί το πρόγραμμα, ενώ είμαστε ήδη στο Δεκέμβριο. Δεν ξέρω πόσο χρόνο ακόμη πρέπει να περιμένουμε ώσπου να υπάρξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να αποτελέσει βάση για πιο ριζικές αλλαγές. Δεν πρόκειται ε, για ε, ευχολόγια, βασιζόμαστε σε αυτό το οποίο προετάθη την, ε, το, πέρυσι. Δηλαδή, είμαστε υπέρ του ΙΤΣ ή του ΣΤΕΤΣ και νομίζω ότι το ΣΤΕΤΣ εδώ προχωρά περισσότερο, χωρίς όμως όλα αυτά τα μέτρα να είναι δραστικά. Οι αλλαγές είναι αρκετά ισοσχελισμένες και η μείωση είναι αρκετά μεγάλη. Δεν νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται χρειάζεται, ε, ότι πρέπει να αγνοήσουμε τα στέξ που είναι επιστημονικές διαπιστώσεις και στις οποίες πρέπει να ε, βασιστούμε. Όσον αφορά την τροπολογία 9, ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα το οποίο να προβλέπει μία αύξηση των ε, επιτρεπτών ε, ημερών αλληλείας αν δεν είναι τόσο μεγάλη η θνησιμότης. Ε, αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο προτείνουμε είναι φυκτό. Το 10% που προτείνουμε δεν είναι υπερβολικό και επιτρέπει να υπάρχει και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα στην ε, ε, Μαύρη Θάλασσα. Τροπολογία 10. Ε, η διατάξεις ε, του άρθρου 8 παράγραφος 6 αναφέρονται στην ε, ε, ελαφρά συγκέντρωση αποθεμάτων γάδου και νομίζω ότι εδώ δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη ότι στα 12 μίλια η κατάσταση είναι διαφορετική. Οπότε θα πρέπει να μπορεί κανείς να, ψηφι... ψαρέψει αυτά τα ψάρια ε, στο χώρο των 12 μιλίων. Και αυτό που μας απασχολεί είναι ότι δεδομένων των διατάξεων κατά τις πέντε ημέρες ε, ε, βασιζόμαστε στα αποθέματα γάδου ε, και τα αποθέματα αυτά διαταράσσονται με το ισχύον σύστημα. Ίσως λοιπόν αυτό το οποίο προτείνω μπορεί να οδηγήσει σε κάποια ισορροπία και δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα την οποία συζητάμε. Ε, δεν χρειάζονται περισσότερες μέρες αλίας. Υπάρχουν δεδομένα ε, όρια. Παραδείγματος χάρη βρισκόμαστε στο 37% Τον ε, ΤΑΚ που προβλέπονται για το τρέχον έτος και που είχαν εξαντληθεί ε, τέλος Σεπτεμβρίου. Οπότε ε, βασιζόμαστε σε συγκεκριμένες ε, διαπιστώσεις και ελπίζω θα μπορέσουμε να το εξετάσουμε και στη συνέχεια. Πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε και περνάμε τώρα το επόμενο θέμα. Τροποποίηση του κανονισμού 1100 για το ευρωπαϊκό χέλι. Η Επιτροπή δεν θα πει τίποτα. Όχι, όχι, έκανα λάθος. Όχι, έκανα λάθος, λέει ο Πρόεδρος. Πρέπει να δω... Εγώ προχώρησα πολύ γρήγορα. Πρέπει να δώσουμε τον ε, λόγο στην Επιτροπή. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν είπατε κι εσείς τίποτα και έτσι έτρεξα κι εγώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε μερικά από τα σχόλια που ακούσαμε όσον αφορά αυτή την έκθεση. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τη γραμματεία καθώς και με τον κύριο Βαλέσα και τη βοηθό του, τους βοηθούς του φέραμε να μελετήσουμε την πρόταση και να μελετήσουμε διάφορες πτυχές και να διευκρινίσουμε πολλά ζητήματα. Κάποια γενικά ζητήματα όταν έχουμε επιστημονικά στοιχεία. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το θέμα είναι ποια επιστημονικά στοιχεία θα λάβουμε υπόψη, λέτε για 12 μίλια. Η εκτίμηση αντικτύπου δεν αναφέρει 12 μίλια, δεν υπάρχει αξιολόγηση τέτοια. Αν κοιτάξετε το χάρτη της Βαλτικής θάλασσας, 12 ε, μίλια, περιοχή 12 μιλίων, αφορά και περιοχές βαθύτερες των 20 μέτρων και είναι περιοχές συνεπώς όπου τοκούν οι γάδοι και θα υπάρχει συνεπώς επίπτωση για τον γάδο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτές τις πτυχές διότι τα σκάφη κάτω των 12 μέτρων εξαιρούνται από ορισμένε απαιτήσει ε, στο πλαίσιο του κανονισμού του Συμβουλίου και αυτή η εξαίρεση είναι πολύ σημαντική. Στην έκθεση λένε ότι ότι εφόσον τηρούνται τα ανώτατα επιτρεπόμενα λιεύματα, τότε μπορούν να παρεκκλίνουν τα σκάφη προς περιοχές βάθους μικρότερου των 20 μέτρων, εφόσον δεν υπάρχει γάδος εάν δούμε το, αυτά τα, 12, τα σκάφη 12 μέτρων και λιγότερα από 12 μίλια θα μπορούσαν να είναι και σε 6 μίλια και σε ορισμένες περιοχές ακόμη και 6 μίλια σε ορισμένες περιοχές των σκανδιναβικών χωρών ε, μπορεί να υπάρχουν βαθύτερα ύδατα στα 6 μίλια και εκεί να διαδράξουμε το ε, γάδο που εκεί. Απλά ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτά τα θέματα και ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και να μελετήσουμε προσεκτικά όλες τις πτυχέ αυτή τη πρότασης. Μια άλλη πτυχή που θα ήθελα να επισημάνω σε αυτή την πρόταση ότι εδώ προτείνουμε παρέκκληση από την θέση που είχε πρωτήτερα υιοθετήσει η Επιτροπή Αλληλείας για τη χρησιμότητα. Μια άλλη πτυχή που προτείνεται και προέκυψε από συζητήσεις όπως έχει αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να συμμορφώνεται αλλά μας ενημέρωσαν ότι ίσως να γίνουν περαιτέρω προσαρμογές στο μέλλον. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανένα ε, συνάδελφος το λόγο. Διαφορετικά θα ολοκληρωθεί το θέμα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θέτουν κάποιες ομάδες σε σχέση με ένα προηγούμενο θέμα. Η ψήφιση της έκθεσης του κυρίου Γκάλαχερ σε σχέση με το πρώτη ε, συμβιβαστική τροπολογία. Λέγουν ότι δεν ψηφίστηκε. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι την ψηφίσαμε. Φαίνεται ότι δεν μπορούμε να κάνουμε επαλήθευση τώρα. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε επαλήθευση, να ψηφίσουμε αφού κάνουμε επαλήθευση, γιατί είμαι σίγουρος. Δεδομένου όμως ότι υπάρχει δυσκολία τεχνική, ας το κάνουμε. Έχω στοιχηματίσει και με τη γραμματεία και θα κερδίσω το στοίχημα και θα φάω... Γιατί θα κερδίσει μεσημεριανό αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας το ξαναψηφίσουμε. Συμβιβαστική τροπολογία 1 της έκθεσης Γκάλαγερ. Την ξαναψηφίζουμε. Είναι θέμα των ομάδων. Τέθηκε το Προεδρείο, εγώ πιστεύω ότι ψηφίστηκε. Ποιος είναι υπέρ, λοιπόν, της συμβιβαστικής τροπολογίας αριθμός 1. Ποιο είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν, περνούμε στο επόμενο θέμα. Σημείο 13. Κανονισμός του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος Ευρωπαϊκού Χελιού. Προηγούμενο θέμα. Τροπολογία κατάθεσης τροπολογιών 15 Οκτωβρίου. Το μεσημέρι. Λήξη της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει το θέμα αυτό, το 13, για την αναστήση στο αποθέμα του Ευρωπαϊκού Χελιού. Έχει το λόγο η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι η τροπή του κανονισμού για την ανασύσταση του αποθέσεων του ευρωπαϊκού χελιού σύμφωνα με τη ΣΛΕ. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής βάσει του κανονισμού άλλαξαν και είναι ε, κατεξου... Ε, ενέργεια, δράση κατεξουσιοδότηση και μέτρα που θα επιτρέψουν να κάνουμε την ασύστηση του στο του Ευρωπαϊκού Χελιού βάσει της σχετικής ε, παραγράφου. Θα πρέπει να δοθεί λοιπόν αυτή η εξισιοδότηση στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 5.1 για να γίνει κάτι τέτοιο. Το παρόν κείμενο του κανονισμού που δίδει στην ε, Επιτροπή ε, αρμοδιότητες για να κάνει τέτοιου είδους, να λάβει τέτοιου είδους μέτρα και να τροπολογήσει κάποια θέματα, είναι δυνατόν, αλλά δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει κατά συνέπεια βάση ε, των ισχυών των άρθρων. Επίσης, συμπληρωματικά, Όσον αφορά τι τροπολογίε ευθυγράμμιση με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, ε, προτείνουμε διάφορε άλλε αλλαγέ σε αυτόν τον κανονισμό. Καθιερώθηκε με αποφασή της Επιτροπής το 2008 ότι η Μαύρη Θάλασσα και τα σχετικά ποταμιά συστήματα δεν αποτελούν φυσικό οικότοπο του Ευρωπαϊκού Χίλιου για τους σκοπούς του κανονισμού. Έτσι λοιπόν το άρθρο 1 παραγράφος 2 του κανονισμού είναι απορχαιωμένο και θα πρέπει να διαγραφεί. Στη συνέχεια, η αίτηση εξαίρεση από την υποχρέωση προετοιμασία σχεδίου διαχείριση ε, του χελιού που πρέπει να κοινοποιηθεί στην Κομισιόν έω την 1η Ιανουαρίου 2008. Η απόφαση του 2009 τη Κομισιόν που εγκρίθηκε από την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Ρουμανία, την Αυστρία και τη Σλοβακία για εξαίρεση από, αυτή την, από αυτόν τον κανονισμό κατά συνέπεια το άρθρο 3 του κανονισμού θα πρέπει επίση να διαγραφεί. Τέλος, επειδή η Κομισιόν δεν κατάφερε να αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα μέτρα που αφορούν την ανασύσταση του πληθυσμού καθώς και την εξέλιξη της τιμής αγοράς μέχρι την 1η Ιουλίου του 2011 λόγω ε, αργής μεταφο... Ε, αποστολής των στοιχείων από τα διάφορα κράτη-μέλη αναβάλει την ημερομηνία για την 31η Δεκεμβρίου του 2012. Οι προτινόμενε τροπολογίε είναι απαραίτητε ώστε ο κανονισμό να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Πιο αργά, παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρο. Κατά συνέπεια, η Κομισιόν ελπίζει ότι η απόφαση θα εγκριθεί εύκολα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ώστε ο κανονισμό να μπορέσει να τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Λέβιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον ο κανονισμός αυτός ο οποίος έρχεται στο Κοινοβούλιο σχετικά με την ε, ε, πολιτική και αντιλαμβανόμαστε ότι τα κράτη-μέλη έχουν μία διαφορετική ε, αντιμετώπιση και δεν είναι αποδεκτή διότι αυτή, αυτός ο κανονισμός του χελιού είχε, είχε καταρτιστεί το 2007. Καταρχήν πρέπει να γνωρίζουμε ότι επρόκειτο για κοινά αποθέματα, δηλαδή υπάρχει ένα είδος μόνος ευρωπαϊκού χελιού και υπάρχει ε, μία εξέλιξη σε τρεις φάσεις. Το ένα είναι ε, το λευκό, το άλλο το κίτρινο και το άλλο το ασημένιο. Ε, και ε, ε, υπάρχει, ε, δεν είναι η κατάσταση η ίδια με τον Σολομό ο οποίος ξεκινά από τα ποτάμια και καταλήγει στη θάλασσα. το χέλι ζει στο, σε νερό και μόνο πηγαίνει για να γεννήσει στη θάλασσα. Κοντά στην περιοχή της ε, της θαλάσσης των Σαργασών και βλέπουμε ότι στη συνέχεια η θάλασσα το χέλι αφού γεννήσει ε, πεθαίνει. Έρχεται στην Ευρώπη με το Gulf Stream. Οπότε ε, πεθαίνει ασχέτως του είδους μετά ε, το, ε, αφού καταθέσει τα αυγά του και όλα τα είδη έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά στο απόθεμα χωρίς να υπάρχουν διαφορετικές 27 φυλές χελιάς και ε, θεωρώ ότι είναι ένα σύμβολο της συνεργασίας και πρέπει να μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκό χέλι, για ένα μόνο είδος και βλέπουμε ότι τώρα εδώ και 20-30 χρόνια τα αποθέματα αυτά έχουν μειωθεί. Από τη δεκαετία του 80 ήδη και το 2003 οι άισις άρχισαν να χτυπάνε καμπανάκια. Εάν δηλαδή δεν ε, δεν μειώσουμε ε, και δεν εξαφανίσουμε ε, την ε, αιτία θανάτου των χελιών που εφείλεται στον άνθρωπο δεν έχουμε μέλλον. Και συνεφωνήθηκε εκείνη την εποχή ένα πρόγραμμα ανάταξης των αποθεμάτων ε, χελιού ε, και αν δεν έχετε τα στοιχεία, εγώ έχετε υπόψη σας ότι τα έχω διαβάσει γιατί είμαι η συγγήτρια για το πρόγραμμα για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού. Υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία διότι λέγεται ότι τα κράτη-μέλη έπρεπε να έχουν υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εθνικά τους προγράμματα ανατάξεως των αποθεμάτων το 2008. Θα ήθελα λοιπόν να, να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσα κράτη ε, είχαν ε, υποβάλει τα προγράμματά τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2008. Το δεύτερον, εφόσον δεν το έπραξαν, αν δεν το έπραξαν, θα έπρεπε να έχουν μειώσει ε, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2009 να έχουν μειώσει την προσπάθεια αλληλείας στο 50%. Πόσοι από αυτοί το έπραξαν ακόμη και αν δεν έστειλαν σχέδια διαχείρισης των αποθεμάτων. Επίσης έπρεπε να στέλνουν ορισμένα στοιχεία που θα επέτρεπαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2011 να αναφερθούν εις ε, τα μέτρα της ε, ε, ανασυστάσεως των αποθεμάτων. Τώρα υπάρχει μία νέα προθεσμία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εφέτος. Έχουμε δώσει δηλαδή ένα, ένα επιπλέον έτος για να κάνουν τη δουλειά που έπρεπε να έχουν κάνει εδώ και καιρό και θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί δηλαδή δεν έχουν υποβάλει τα στοιχεία τα οποία έπρεπε να έχουν υποβάλει για να επιτρέψουν στην Επιτροπή να ενημερώσει το Συμβούλιο. Αυτά Επίσης, το τρίτο βήμα είναι ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να προβούν σε μία αξιολόγηση των διαφόρων εθνικών προγραμμάτων και να την υποβάλουν μέχρι το καλοκαίρι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσα από τα κράτη το έπραξαν και στη συνέχεια ερχόμαστε στον κανονισμό και στους στόχους του κανονισμού μελέτησα πολύ προσεκτικά την ε, ε, γνωμοδότηση της ΆΙΣΙΣ η οποία άρχισε να λέει εδώ και χρόνια ότι η ανασύσταση των αποθεμάτων του χελιού δηλαδή ε, εάν έπαιρναν αποθέματα από την Νότιο Ευρώπη χελιού και τα τοποθετούσαν στη Βόρειο Θάλασσα παραδείγματος χάρη δεν θα ήταν μία μία σωστή λύση σύμφωνα με την ΆΙΣΙΣ η οποία επανέλαβε πέρυσι ότι αυτό δεν θα βοηθήσει στην ανασύσταση του αποθέματος και λένε στη συνέχεια επιπλέον στην έκθεση αυτή ότι χρειάζονται ε, πολύ περισσότερες προσπάθειες για να επιβιώσει το απόθεμα του ευρωπαϊκού χελιού διότι εάν παίρνετε ένα χέλι από την ε, ε, ε, στην ε, Νότιο Ευρώπη ε, για να φτάσουν ε, και να προσαρμοστούν στη Βαλτική και να γίνουν κίτρινα χέλια παραδείγματο χάρη μετά από 20 χρόνια που θα έχουν αποκατασταθεί τα αποθέματα θα ξαναφύγουν προς την θάλασσα των Σαργασών για να υπάρχει οτοκία και για το λόγο αυτό αναρωτιέμαι αναρωτιέμαι τι μπορεί να γίνει. Είναι ένα από τα μέτρα που επιτρέπονται εις ε, την ε, Ευρω... ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό για να υπάρξει ανασύσταση ε, των αποθεμάτων. Αλλά δεν θα επιτρεφθεί αυτό διότι δεν μπορεί κανείς τέχνητα για να επιβιώσει ή βιομηχανία αλίας των χελιών να υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα και τα τα Πρέπει να υπάρξει μία αξιολόγηση, πράγμα που έχει γίνει παραδείγματο χάρη ή στην Σουηδία, η οποία παρόλο που βασίζεται στα αποθέματα του χελιού, έχει μειώσει 50% την αλληλεία, ε, απέχει πολύ από το να επιτύχει το στόχο του κανονισμού που είναι 40% ε, ε, διαφυγή των χελιών που έχουν μεγαλώσει ε, σε ελεύθερο περιβάλλον. Παρόλο που αυτό μας φαίνεται, μας φαίνεται πάρα πολύ θεωρητικό. Το μόνο μέτρο λοιπόν το οποίο ε, έχει βρεθεί είναι να σταματήσει στην Ιρλανδία παραδείγματο χάρη τελείω η αλληλεία του χελιού. Και βλέπω ότι στην αξιολόγηση ούτε η Ιρλανδία πετυχαίνει το στόχο που είχε θέσει. Άρα δεν μπορούμε ε, να εξασφαλίσουμε ότι 40% του ελεύθερου πληθυσμού θα επιβιώσει. Και ε, έρχομαι εδώ ε, στην ανάγνωση της πρώτης γραμμής της γνωμοδότησης της ISIS για το χέλι το 2012 όπου λέει ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη και χρειάζεται επίγουσα δράση και ε, πρέπει να διαγραφεί η ανθρωπογενής θνησιμότητα η οποία επηρεάζει την παραγωγή και θα πρέπει ε, η θνησιμότητα να φτάσει στο 0% μέχρι ότου διαπιστωθεί ότι αυξάνονται τα αποθέματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, υπάρχει ένας κύκλος και Αυτός ισχύει εδώ και δύο εκατομμύρια χρόνια ε, ακολούθησε τις κινήσεις της τεκτονικής πλάκας και έτσι βρέθηκε στη θάλασσα των Σαργασών και τώρα βλέπουμε ότι αυτό το αρχαίο ζώο εξαφανίζεται και πιστεύω ότι είναι μεγάλη ανησυχία και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Πέραν αυτού θέλω να, ρωτήσω, ε, ε, να θέσω μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι δεν την παρουσίασε ε, προηγουμένως διότι μιλάτε για το άρθρο 9 παράγραφος 3 όπου τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επέμβουν με τις ε, μελέτες αξιολογήσεως και λέτε στην παράγραφο αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει αυτών των στοιχείων θα προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για να επιτευχθεί με μεγάλη πιθανότητα ο στόχος της ανασύστασης του αποθέματος του χελιού και δεν καταλαβαίνω γιατί εσείς διαγράφετε όλη την παράγραφο. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι όταν τα κράτη έχουν υποβάλει τα προγράμματά τους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει και αν δεν επιτευχθεί ο στόχος τότε η Επιτροπή θα πρέπει να διατυπώσει μία νέα πρόταση και δεν καταλαβαίνω γιατί το διαγράφεται από αυτό το σημείο. Η γενική άποψη της Επιτροπής η εντύπωση η οποία δίδεται εφόσον είχατε τη δυνατότητα να εξετάσετε την αξιολόγηση των κρατών μελών που υπευλήθη φέτος το καλοκαίρι ε, για να προχωρήσουμε στην επίτευξη του στόχου ο οποίος δεν εξασφαλίζεται από την ISIS και σύμφωνα με την ΆΙΣΙΣ τουλάχιστον 50% θα επαρκούσε. Ε, αυτές είναι οι τροπολογίες που έχω. Ευχαριστώ. Ένας μόνο συνάδελφος μου στο λόγο, δεν ζητάει κανείς άλλος. Για να υπολογίσει το χρόνο το λέω, ο κύριος Ντέιβις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέχθη ότι 99% των αποθεμάτων έχουν καταστραφεί. Δεν ξέρω ποιο δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει. Η συγγήτρια η Κομισιόν. Δεδομένου λοιπόν ότι ακούσαμε πως έχουν σήμερα τα ε, αποθέματα του ευρωπαϊκού χελιού, ίσως να είναι 99,9 κατεστραμμένα. Υπάρχει πουθενά κανένα σημείο αισιοδοξία. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ για όλε τι παρατηρήσει και τι ερωτήσει σα Πριν δώσω το λόγο στον τεχνικό μα εμπειρογνώμονα, θα ήθελα να τονίσω απλά ότι ο κανονισμό αυτό ε, σκοπό ουσιαστικά τη πρόταση τη Κομισιόν είναι η ευθυγράμμιση του κανονισμού με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Γι' αυτό το λόγο επικεντρωθήκαμε στην αναταξινόμηση των εξουσιών και εκαθαρίσαμε κάπως τον κανονισμό. Δεν προχωρήσαμε περαιτέρω σε αναθεώρηση όλου του κανονισμού και του περιεχομένου του. Τώρα όσον αφορά την ερώτηση για το άρθρο 9 παραγραφος 3 και το δικαίωμα της Κομισιόν να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα πράγματι διαγράφηκε διότι σκοπός ε, ήταν να προτείνει μέτρα η Κομισιόν τα οποία στη συνέχεια θα αποφασίζονται από το Συμβούλιο ε, η διαγραφή λοιπόν αυτής της παραγράφου σημαίνει απλά ότι η Κομισιόν διατηρεί το δικαίωμα πρωτοβουλίας του όπως προβλέπεται στη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το άρθρο 17 και ανά πάσα στιγμή που το θεωρεί ε, σκόπιμο μπορεί να προτείνει κατάλληλα μέτρα. Όχι μέσω κατεξουσιοδότηση εκτελεστικών πράξεων, αλλά μέσω τροποποίησης του κανονισμού και διαδικασία συναπόφασης. Ευχαριστώ. προσθέσετε κάτι, κύριε Συγγνώμη, συγγνώμη, να ακούσουμε την Κομισιόν ακόμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ίσως να απαντήσω σε τρία σημεία. Επειδή τα τεχνικά σημεία που αναφέρθηκαν από την κυρία Λέβεν είναι συναρπαστικά, εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Θα μπορούσαμε να περάσουμε πολλέ μέρε να τα συζητάμε. Πολύ ευχαριστώ, το έκανα, αλλά δεν έχουμε τόσο χρόνο αυτή τη στιγμή για να συζητήσουμε τι τεχνικέ πτυχέ. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω τα εξή. Πρώτον, όσον αφορά τι καθυστερήσει σε ορισμένε από τι προθεσμίε που αναφέρατε, ξεκινήσαμε με την πρώτη προθεσμία που ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2008, προθεσμία δηλαδή για την υποβολή των σχεδίων διαχείρισης των κρατών μελών στην Κομισιόν. Σημειώθηκαν κάποιες καθυστερήσεις, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ποιος ε, υπέβαλε το σχέδιο και πότε. Υπήρξαν καθυστερήσεις λοιπόν λόγω της εξαιρετικά τεχνικής και πολύπλοκης φύσης αυτού του κανονισμού. Οφείλονται επίση οι καθυστερήσει στο γεγονό ότι πολλά από τα σχέδια, ουσιαστικά η πλειοψηφία του, ίσω μία δύο εξαιρέσει, χρειάστηκε να αξιολογηθούν και να επανασταλούν στα κράτη-μέλη, ώστε αυτά να παρέχουν περισσότερε διευκρινήσει, πληροφορίε και ξανά πίσω στην Κομισιόν και τελικά στην ISIS για την τεχνική αξιολόγηση. Αυτή η αρχική καθυστέρηση λοιπόν οδήγησε και σε καθυστέρηση εφαρμογής των σχεδίων καθώς και σε καθυστέρηση της υλοποίησης των μέτρων ανασύστασης του πληθυσμού διότι δεν είχαμε λάβει τις τιμές που καταβλήθηκαν για την ανασύσταση και έτσι καθυστερήσει και η έκθεση τιμολόγηση. Τώρα για να απαντήσω στον κύριο Ντέιβις όσον αφορά το 99 ή το 99,9% αυτή τη μείωση που αναφέρθηκε ε, του αποθέματος αυτό το ποσοστό συχνά ε, σχετίζεται με τη μείωση των νέων χελιών ουσιαστικά που έρχονται από τη θάλασσα των Σαργασών δεν αφορά μείωση του τρέχοντος αποθέματος που, που, ζει στα ευρωπαϊκά ύδατα. Τέλος, κατά πόσο μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Καλή ερώτηση. Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε κάποια τάση. Έχουμε τις πρώτες εκθέσεις πρόοδο από τα κράτη-μέλη που καλύπτουν περίπου δύο χρόνια υλοποίηση των σχεδίων. Ωστόσο, μια γενιά χελιών να χρειάζεται περίπου 5 με 20 χρόνια. Μπορεί να χρειαστούν δηλαδή μέχρι 20 χρόνια μέχρι να οτοκίσουν και να οριμάσουν. Και ίσως χρειαστούν δύο ή τρεις γενιές πριν μπορέσουμε να ε, προσδιορίσουμε κάποια συγκεκριμένη τάση. Συνεπώς δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι ακόμη. Ευχαριστώ. Κύριε εντάξει. Σας ευχαριστώ για αυτή τη διευκρίνηση. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Κάποια κράτη-μέλη ε, δεν υποβάλλουν σχέδια, γιατί είναι πάρα πολύ τεχνικά. Και πριν όμως ε, να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός, συζητούσαν για πέντε χρόνια και είχαν ένα μισή χρόνο για να υποβάλουν τα δικά του σχέδια. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, ένα κράτο μέλος που δεν έχει υποβάλει το σχέδιο στην Κομισιό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008 προς έγκριση ή θα πρέπει να μειώσει τις προσπάθειες ελίας ε, κατά ποσοστό 50% σχέση με αυτά που ίσχυαν προηγουμένως ή να τα μειώσει και να ε, σε ποσοστό ε, επίσης, κατά 50% η μείωση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2009. Αυτό ωραίο μου φαίνεται και είναι κάτι το οποίο όλοι θα θέλαμε να το συμπεριλάβουμε σε όλα τα περιφερειακά σχέδια τα αναπτυξιακά για να πούμε δεν το κάνετε όλοι σας δεν θα είναι καλά τα πράγματα δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει καμία εξουσία η Κομισιό. Δεν μπορεί να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη ή να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν ή να κάνει τη μία στο 50%. Γιατί δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Είναι τρομερό αυτό, είναι φανταστικό. Τι μάθημα μαθαίνουμε από εδώ. Κάποιος τρόπος θα πρέπει να υπάρχει. Εάν ε, λοιπόν ε, αναθέτουμε αρμοδιότητες και δεν κάνουμε τίποτε, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι, δεν κάνουν, ότι τα κράτη-μέλη δεν κάνουν τίποτα και συνεχίζουν, εμείς συνεχίζουμε εδώ το μπλα μπλα. Μετά από την ερώτηση του κυρίου Ντέβιση, με την συμφουλή του κυρίου Άισις, το Glass Hill, αυτό το to 1979 average in the Atlantic region and to less ε, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που έχω εγώ και τη μείωση σε ποσοστό ε, λιγότερο από 1% σήμερα με αυτά που λέει η ISIS λοιπόν δεν βλέπω καμία αισιοδοξία να διαγράφεται για το μέλλον. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ η Κομισιό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Απλώς για να απαντήσω σε αυτό το οποίο ελέγχθη για την κύρωση του 50%. Δεν θέλω να ονοματίσω κανέναν. Υπάρχουν όμως δύο κράτη-μέλη τα οποία εφαρμόζουν αυτό το 50%, αντιμετωπίζουν αυτό το 50%, πρέπει να το εφαρμόσουν μάλλον, διότι δεν υπέβαλαν τα σχέδια τους. Άρα τώρα έχουν, ε, πρέπει να έχουν μείωση 50%, τουλάχιστον έχουμε μία περίπτωση άλλης χώρας που είχε μία μικρή καθυστέρηση όσον αφορά την ε, υποβολή των σχεδίων και πάγωσε τα πράγματα η Κομισιό μέχρι να υποβληθεί αυτό το σχέδιο Ναι, κύριε Λέβεν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω λάβει εγώ, ένα κράτος που έχει μειώσει την προσπαθία της είναι η Βουλγαρία, αλλά εξαιρείται γιατί είναι μαύρη θάλασσα. Μου κάνετε νόημα τώρα. Η Κομισιόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. μέρος του εδάφους της Βουλγαρίας βρίσκεται στη λεκάνη το Δούναβη και μέρος εκτός ορισμένα δηλαδή από τα ποτάμια της Βουλγαρίας ε, καταλήγουν στο Αιγαίο και ένα κομμάτι του Δούναβη βρίσκεται στο εδαφός της η εξαίρεση αφορά το κομμάτι που βρίσκεται στο Δούναβη έχουν μια εξαίρεση δηλαδή στο κομμάτι του εδάφους τη ε, που βρίσκεται στη λεκανή του Δούναβη. Για εκεί δεν χρειάζεται να υποβάλουν σχέδιο, αλλά υποτίθεται ότι έπρεπε να υποβάλουν σχέδια για τα ποτάμια συστήματα που καταλήγουν στη Μεσόγειο, στη, στο Αιγαίο. Δεν υπέβαλαν τέτοια σχέδια και έτσι υφίστανται κυρώσει σε σχέση με την Αλία σε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Διακόπτουμε τη συνεδρία σας. Ευχαριστούμε καθώς και τους τερμηνείς. Στις 3 ακριβώς θα ξαναγυρίσουμε εδώ σήμερα το απόγευμα. Γεια σας.